Έχετε το λόγο κύριε Παρβανό για πέντε λεπτά. Κυρία Παρβάνοβα. Dear President, dear Madam Commissioner. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους σκιώδει εισηγητές, το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών και την Οργάνωση για την Υποστήριξη των Θυμάτων για τη συνεισφορά τους στην έκθεση αυτή. Η βία κατά των γυναικών είναι σημαντική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια μορφή διακριτική μεταχείρισης που βασίζεται στι ε, διαφορέ των φύλων και δεν επιτρέπει στις γυναίκες να συμμετάσχουν πλήρως ε, στην οικονομική και πολιτική και κοινωνική ζωή. Ε, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, ε, περίπου 20-25% των γυναικών στην Ευρώπη έχουν τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή τους υποστεί βία και περίπου 10% έχουν υποστεί σεξουαλική βία. 12 με 15% των γυναικών στην Ευρώπη είναι θύματα ε, οικογενειακής βίας ε, και ε, υπάρχουν πολλοί θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της οικογενειακής βίας. 220 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο υπολογίστηκαν το 2011 οι ζημίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιχειρήσεις, για τις υπηρεσίες και επίσης και από το κόστος των τραυμάτων της βίας έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή να διαμορφώσουν μια νέα ευρύτερη στρατηγική και νομοθεσία για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια νομοθετική πράξη που να δημιουργεί το υπόβαθρο για να προστατεύονται οι γυναίκε, ούτε υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Το επίπεδο προστασία των γυναικών και των κοριτσιών στα 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ποικίλει κατά πολύ. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα διασυνοριακό πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κοινοί ορισμοί και κάποια ελάχιστα πρότυπα. Στην έκθεση περιλαμβάνεται και ένα ψήφισμα και στο παράρτημα ε, βασίζεται στο άρθρο 84 της Συνθήκης για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής και εκπαίδευση των εμπλεκομένων ε, υπαλλήλων και στο άρθρο 83α της συνθήκης υπάρχει βάση για μια τέτοια δράση σχετικά με το διασυνοριακό χαρακτήρα τέτοιων μέτρων. Μέχρι το τέλος του 2014 θα πρέπει να υποβάλουμε μια πρόταση για μέτρα των κρατών μελών για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Ακόμη ε, θέλουμε να έχουμε ένα ε, σύστημα συλλογής στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και ζητάμε από την Επιτροπή να ε, διαμορφώσει ένα σχέδιο που θα ασχολείται με την πρόληψη ε, της βίας κατά των γυναικών. Ζητάμε από την Επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία για να ε, προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση κατά της βίας. Ζητάμε ακόμη να υποστηριχθούν τα ε, μέσα και οι φορείς που ασχολούνται με τη βία των γυναικών και η Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει αυτά τα μέτρα σε διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει ότι όλες οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να ζουν χωρίς προβλήματα βίας εναντίον τους. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να ψηφίσουμε την ε, έκθεση αυτή και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να δεσμευθεί στεναρά υπέρ αυτών των μέτρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Παραβάνοβα. Έχουμε τώρα τη διαδικασία KFCI. Περισσότερες αιτήσει από ό,τι προβλεπόμασταν και δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πέντε λεπτά. Δίνω καταρχήν το λόγο στην κυρία Αντζελίδη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια δυστυχώς επιβεβαιούνται πάντα τα ίδια δραματικά δεδομένα. Μία γυναίκα στις τέσσερις έχει υποστεί βία έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής της και 10% σεξουαλική βία. Η καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών θα πρέπει να καταστεί μια πραγματική προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η μηδενική ανοχή. Ζητάμε να υπάρξει μια οδηγία γι' αυτό, γιατί η βία εις βάρος των γυναικών είναι ένα σοβαρότατο έγκλημα. Απαιτείται μια οδηγία για τον καθορισμό αυστηρών νόμων, αποτρεπτικών, που να ισχύουν και στις 28 χώρες της Ένωσης. Απαιτείται επίσης και ένα ισχυρό πρόγραμμα δράσης για ενημέρωση και πρόληψη στην καταπολέμηση της βίας. Ευχαριστώ κύριε κύριε Πρόεδρε. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι απίστευτο να μην υπάρχει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Μία από τις τέσσερις γυναίκες έχει υποστεί την βία αυτή έστω και μία φορά και 10% έχουν υποστεί σεξουαλικές μορφές βίας. Αυτό δεν είναι κάτι που εκφράζεται μόνο με αριθμούς, γιατί φοβάμαι ότι οι στατιστικές μεθοδολογίες που ακολουθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι ικανοποιητικές. Ξέρουμε ότι το 1,8 του ΑΕΠ δαπανάται για την αντιμετώπιση σε ιατρικό και νοσοκομιακό επίπεδο των συνεπειών αυτής της μορφής βίας. Είναι καθήκον μας λοιπόν να προστατεύσουμε το μισό του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από 3.000 γυναίκε πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη σαν αποτέλεσμα βία εναντίον του λόγω φύλου. Πολλά κράτη-μέλη δεν κρατάνε στατιστικέ για τα θέματα αυτά, θεωρούν ότι είναι ένα οικογενειακό θέμα, ένα οικιακό θέμα η βία αυτή η ενδοοικιακή. Η, η διάσταση αυτού του προβλήματο είναι τεράστια και αποτελεί μια μορφή περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρώπη. Θέλουμε μια πολιτική η οποία να βασίζεται στην προστασία των ε, θυμάτων, στη δίωξη αυτών των αδικημάτων και ιδίω στην πρόληψή του. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη μάστιγα η οποία πρέπει να εξαλειφθεί με επιμονή στις αξίες και στην πρόληψη. Θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε καλύτερη συμβίωση και μια μορφή, που θα, μια μορφή συμβίωση που θα αποτρέψει τη βία κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόμασιτς. Kao žena i bivša dugogodišnja policijska službenica posebno sam zainteresirana za rješenje ovog problema te dajem otvorenu podršku borbi ως γυναίκα και πρώην αστυνομικός ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Υποστηρίζω το ψήφισμα αυτό ιδίω το να υπάρχουν προληπτικά μέτρα και μέτρα ευαισθητοποίησης των πολιτών για το πρόβλημα αυτό. Πιστεύω ότι τέτοιες εκστρατείε θα πρέπει να αποτελούν τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος και θα πρέπει να προσφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την καριέρα μου ως αστυνομικός έχω δουλέψει και με γυναίκες θύματα βίας και γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα μας αρκέσει το απλώς να ψηφίσουμε νομοθετικά κείμενα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών στο δρόμο, ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους και όχι μόνο στους διαδρόμους των Βρυξελών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τοπικές ιδιομορφίες και τα κράτη-μέλη έχουν περισσότερες αρμοδιότητες σε αυτό το τομέα από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ την κυρία Τόμασιτς και κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Στη Ρουμανία ε, υπάρχει μεγάλο ποσοστό οικογενειακής βίας ε, και μία στις τρεις γυναίκες ε, είναι θύμα οικογενειακής βίας. Η βία κατά των γυναικών είναι μια σκληρή πραγματικότητα και αυξάνονται τα σχετικά κρούσματα. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της ε, Ρουμανίας συνεχώς αναβάλει την ε, επικύρωση του πρωτοκόλου της Κωνσταντινούπολης ε, και δεν θα πρέπει να υπάρχει καθόλου ανοχή για τέτοιες υποθέσεις βίας κατά των γυναικών. Σε πολλές περιπτώσεις η συμπεριφορά προκύπτει από την ε, εκπαίδευση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραμελούμε σημαντικά στοιχεία. Τα παιδιά του σήμερα, οι ενήλικοι του αύριο, θα συμπεριφέρονται όπως τα έχουμε εκπαιδεύσει στην οικογένεια και στο σχολείο. Κυρία Λουπτσεβά. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτικά διαστήματα εξετάζει εκθέσεις σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών, δυστυχώς. Το θέμα αυτό δεν έχει βρει μια επαρκή λύση. Η βία κατά των γυναικών είναι μια έκφραση Σκέψεις και συμπεριφοράς που προκύπτει από την ανισότητα των δύο φύλων. Οδηγεί σε σωματική ταλαιπωρία και των θυμάτων αλλά και των οικογενειών τους και περαιτέρω οι θύτες μένουν ατιμόρυτοι. Δεν χρειάζεται μονάχα ε, νομική υποστήριξη αλλά και ψυχολογική και κοινωνική βοήθεια για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα τραύματα αυτής της κακοποίησής τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά που γίνονται θύματα αυτής της βίας απαιτούν προσπάθειες για να υπάρξει η σωστή πρόληψη αυτών των ενεργειών. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα πρέπει να είναι πιο ενεργό στον τομέα αυτό και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκέ ρυθμίσει για τα θέματα αυτά και καλύτερη πληροφορία και κατάρτιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λιούψεβα. Είπα δεν μπορώ να δώσω σε όλους το λόγο και υπήρξα αρκετά ε, γενναιόδωρος ήδη. Έδωσα σε πολλούς το λόγο στη διαδικασία ΚΑΣΤΙΑ και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Γιώργεβα, την Επίτροπο κυρία Γιώργεβα για την λήξη της συζήτησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε καθημερινή βάση οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες υφίστανται επιθέσεις, μειώνεται η αξιοπρέπειά τους, τραυματίζονται, πεθαίνουν μερικές φορές μόνο και μόνο γιατί είναι γυναίκες και κορίτσια. Και αυτό συμβαίνει και στα κράτη-μέλη, συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Επηρεάζει φυσικά τις γυναίκες που είναι θύματα, αλλά και είναι και ένα τεράστιο πρόβλημα για το σύνολο της κοινωνίας. Είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ την κυρία Παρβάνοβα, να την ευχαριστήσω για την έκθεσή της, να υπογραμμίσω τον αγώνα τον οποίο δίδει εναντίον της βίας εις βάρος των γυναικών και για την έκκλησή της να την ευχαριστήσω επίσης ε, για δράση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς δείξαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των κοινοτικών αρμοδιοτήτων για να προλάβουμε και να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές βίας και εις βάρος των γυναικών στην καθημερινή μας σχέση και με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό το υπογραμμίζω και στον δικό μου τομέα, τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε ένα συνολικότερο πλαίσιο νομικό, θεσμικό για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Περιλαμβάνουμε εδώ την οδηγία για την καταπολέμηση του τράφικινγκ ανθρωπίνων όντων, την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, τον κανονισμό για θέματα που αφορούν την αστική πλευρά των διώξεων, όπως επίσης και τα δικαιώματα των γυναικών, υπογραμμίζοντας την μεγάλη ανάγκη που έχουν τα θύματα βίας για φιλετικούς λόγους. Έχει υπάρξει λοιπόν ένα πλαίσιο νομικό, καθοδηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σωστή εφαρμογή στα κράτη-μέλη αυτής της νομοθετικής ρύθμισης. Όπως προτείνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν δυνατότητες για πιο φιλόδοξες ρυθμίσεις, κάτι το οποίο προαπαιτεί βέβαια μια προσεκτική ανάλυση για το τι ε, ε, μπορεί να γίνει στα πλαίσια της κατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το άρθρο 84 της Συνθήκης της Λισαβόνας θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς για την εναρμόνιση των ποινικών εθνικών ρυθμίσεων στα πλαίσια των κανονισμών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πιθανότητα θετικής προστιθέμενης αξίας και τέτοια πρωτοβουλία. Πρέπει όμως να αξιολογηθεί αυτό από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη πάρα πολλές δραστηριότητες, ανταλλαγές εμπειριών, χρηματοδότησης εκστρατιών ευαισθητοποίηση και δραστηριοτήτων πρόληψης της βίας εις βάρος των γυναικών. Παρ' όλα αυτά συμφωνώ μαζί σας κυρία Παρβάνοβα, πρέπει να βελτιώσουμε τις γνώσεις που έχουμε στον τομέα αυτό και πρέπει οι γνώσεις αυτές να γίνουν δράση και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο κοινοτικό. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχουμε δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό και στα πλαίσια του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και στα πλαίσια της Υπηρεσίας για τον Σεβασμό των Προσωπικών Δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει την σωστή εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών από πλευράς των κρατών μελών. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης και το νέο πρόγραμμα ισότητας για την στήριξη των προσπαθειών που τίνουν στην ανταλλαγή χρηστών πρακτικών και την ενίσχυση των ΜΚΟ που εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα. Η Επιτροπή υιοθέτησε επίσης πρόσφατα και ε, για μέτρα για την καταπολέμηση της ε, κλειτοριδεκτομής και έχει οριστεί και μία μέρα ε, για την ημέρα μηδενικής ανοχής απέναντι στο απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ε, σαν στόχο την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών και της οικιακής βίας και κοιτάμε να δούμε και σε ποιο βαθμό υπάρχουν κοινοτικέ αρμοδιότητας και σε σχέση με τις διεθνείς συμβάσεις. Πάντως το σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να υπογράψουν και να υποκυρώσουν την σύμβαση αυτή. 20 χώρες έχουν υπογράψει αλλά μόνο 3 έχουν επικυρώσει η Αυστρία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Για όλους εμάς εδώ λοιπόν που δεν είμαστε Ιταλοί, Αυστριακοί ή Πορτογάλοι, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να πιέσουμε τα κοινοβούλια των χωρών μας και τις κυβερνήσεις μας, γιατί τα, τα μέσα ενημέρωσης διαρωτώνται γιατί δεν έχουν επικυρώσει τα κράτη-μέλη το μόνο και πρώτο διεθνές μέσο για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Φοβούνται κάτι. Μπορούν να εργαστούν τα νομικά συστήματα προστασίας στις χώρες μας. Και τότε γιατί δεν επικυρώνουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Απαιτούμε πρόοδο λοιπόν και ελπίζουμε να υπάρξει σύντομα στον συγκεκριμένο αυτό τομέα. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόσει τις δυνατότητες που έχει το θέμα δεν είναι μόνο η ισότητα, το θέμα είναι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και προστασία των γυναικών από την βία προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Ευχαριστώ κυρία Τζόρτζεβα. Κλείνει η συζήτηση για το σημείο αυτό. Η ψηφοφορία θα είναι αύριο το μεσημέρι στις 12. Περνάμε στην έκθεση Hannibal, σεξουαλική εκμετάλλευση και πορνεία και ο αντίκτυπό του στην ισότητα των φίλων. Η συγκίτρια έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ του συναδέλφου και ιδίω όλου του σκιώδεις συγκίτρια.